President. Eine Minute. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich erkläre die Κυρίες και κύριοι, ξαναρχίζει η Σύνοδος της Ολομέλειας σχετικά